Ε, απόφαση. Ο κύριο ε, Μπορέλη εγκατέλειψε το EFTD από το 13 2018 και τώρα ανήκει στου μη εγγεγραμμένου. Η κυρία Ρίκελ Ζεκάλσον εγκατέλειψε το ECR από 21η Δευτέρου του 2018 και τώρα ε, ανήκει στου μη εγγεγραμμένου. Η κυρία Γκέρλινγκ εγκατέλειψε το ECR και προσεχώρησε στο ΕΛΚΑ από 28 Δευτέρου του 2018. Ο κύριο Άσουαρτ εγκατέλειψε το ΕΣΥΑΡ και προσχώρησε το ΕΣΤΟΕΛΚ από 28 Δευτέρου του 2018. Ho ricevuto dal gruppo del Partito Popolare Europeo la richiesta di nominare Το ΕΛΚ έχει ζητηθεί ο ορισμό του κυρίου Ντιντιέ ω μέλο αντιπροσωπεία για σχέση.